Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, το 2010 ο Γέρζι Μπούζεκ δήλωσε μαζί με τον Ζακ Ντελόρ και παραθέτω Χρειαζόμαστε ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε την ενέργεια. Είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή και πιο δυνατή ενεργειακή πολιτική. Στις, ε, στους πολιτικούς προσανατολισμούς του, ο ε, νέος πρόεδρος Jean-Claude ε, βασίστηκε σε, αυτήν, σε αυτό το όραμα έτσι ώστε να αναφέρει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι πιο ανεκτική, ανθεκτική συγγνώμη, όσον αφορά την ενέργεια και να έχει ε, πολιτική ελπιδοφόρα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Ε, στο Lettre που μου απίφθινε ε, μου Je suis très fier. Με υπό την ένταση βεβαίως της δικιάς σας σύμφωνης γνώμης να ασχοληθώ με τα θέματα αυτά. Είμαι, είναι τιμή και χαρά ε, για, που μου απέφθηνε αυτή την ε, Οι πολιτικές ενέργεια και κλιματικής αλλαγής ε, βεβαίως βρίσκονται στις, πρώτε πρώτες τη πολιτική πολιτικής ατζέντα. Σήμερα η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει δύο άμεσε ενεργικές προκλήσει. Πρώτα απ' όλα ε, να ε, διασφαλίσει διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια, κυρίω στα πλαίσια τη κρίση μεταξύ τη Ρωσία και τη Ουκρανίας, ενώ από την άλλη πλευρά θα πρέπει να ε, καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ. στην προηγούμενη μακρόαση τόνισα ότι έχουν περάσει 25 χρόνια από την κατάρρευση του σιδερού παραπετάσματος και 10 χρόνια από την ε, προσχώρηση της χώρας μου και των χωρών της Κεντροανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έδωσε τέλος στον τεχνητό αυτό χωρισμό της Ευρώπης. Είναι σημαντικό λοιπόν να σκεφτούμε τη σημασία της δημιουργίας μιας ενεργειακής υποδομής αυτή είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει μονάχα την οικονομική θεώρηση. Με τα γεγονότα των τελευταίων ετών φαίνεται ότι είναι μια τεράστια προτεραιότητα σε επίπεδο στρατηγικής και ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό το θέμα θα είναι μια πραγματική προτεραιότητα για μένα και θα το αναλάβω με, μεγάλη, με μεγάλο αίσθημα ευθύνη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι ε, και εγώ ήμουνα Υποψήφιο σε ευρωεκλογέ και εξελέγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουν τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, να μπορούν οι πολίτες να έχουν θέσει εργασία, να μπορούν να έχουν οικονομική ανάπτυξη και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε πλήρως την πιο δύσκολη κρίση που πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τους πολίτες μας είναι το θέμα των ενεργειακών τιμών. Ο χειμώνα του 2009 είναι ένα χειμώνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ γιατί η Σλοβακία ουσιαστικά βυθίστηκε στο σκοτάδι. Για πάνω από δύο εβδομάδε δεν λειτουργούσε η οικονομία. Μόνο τα νοσοκομεία και τα νοικοκυριά είχαν ενέργεια ενώ είχαν κλείσει τα εργοστάσια. Ξέρετε βέβαια ότι δεν ήταν η μοναδική χώρα η Σλοβακία σε αυτή την κατάσταση χωρί την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την άμεση ευρωπαϊκή αρρωγή. Οι συνέπειε αυτόν το γεγονότο θα μπορούσαν να είναι πραγματικά φρικτές. Γι' αυτό είναι το πραγματικό μας καθήκον, το επιτακτικό μας καθήκον να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας θα αντιμετωπίσουν και πάλι τέτοιες καταστάσεις. Είναι σημαντικό το ότι έχουμε αντλήσει διδάγματα από αυτή την κρίση. Όπως έδειξαν οι δοκιμασίες αντοχής για το φυσικό αέριο, είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε την Ουκρανία με ανάδρομη ροή φυσικού αερίου από τη Σλοβακία, την Πολωνία και την Ουγγαρία. Και αυτό είναι πολύ σωστό γιατί βλέπουμε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί την παροχή φυσικού αερίου σαν όπλο άσκηση πίεση και ω πολιτικό όπλο εναντίον τη Ουκρανία και άλλων χωρών που θέλουν να βοηθήσουν την Ουκρανία. Αυτό είναι απόλυτα παράδεκτο. Εάν αποκομίσω την υποστήριξή σα, θα αντιμετωπίσω το θέμα τη ενεργειακή ασφάλεια και θα του δώσω την πρωταρχική προσοχή μου, λαμβάνοντας υπόψη το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. <clears throat> Οι δοκιμασίες αντοχής έδειξαν ότι μπορεί να περιοριστεί ο αντίκτυπος μιας μείωσης της ροής ε, φυσικού αερίου αν εργαστούμε όλοι από κοινού και δεν έχουμε καθαρά εθνικές προσεγγίσεις. Έχει έρθει η χρονική στιγμή για μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Για αυτού οι οποίοι είχαν σκεπτικισμό για τα θέματα αυτά, θα του θυμίσω ότι πριν από 70 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν απλώ ένα όνειρο. Ήταν αδιανόητο πριν από 25 χρόνια να περάσει κανεί τα σύνορα από τη Σλοβακία στην Αυστρία. Μια τραπεζική ή νομισματική ένωση θεωρείται ότι ήταν κάτι το απόλυτα μη ρεαλιστικό. Όπω είπε ο Νέλσον Μαντέλα, όλα φαίνονται ότι δεν είναι εφικτά μέχρι κάποιο να τα κάνει. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει για να έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Θέλω μαζί σας και τα κρατη να οικοδομήσουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση Ενέργειας που να βασίζεται σε πέντε πυλώνες. Πρώτα απ' όλα <clears throat> η ασφάλεια, η αλληλεγγύη και η εμπιστοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κύρια αγορά ενέργειας με μισό δισεκατομμύριο καταναλωτές. 53% της ενέργειάς μας είναι εισαγόμενη σε κόστος 400 δισεκατομμυρίων το χρόνο. Είμαστε ο μεγαλύτερο ενεργειακός πελάτης στον χώρο, στον πλανήτη μας. Το δείχνουμε όμω αυτό. Έχουμε την ικανότητα να πιέσουμε για να έχουμε δίκαια αντίτιμα για την ενέργεια και καλύτερες συνδικές αγορέ. Σίγουρα όχι. Η έλλειψη ικανότητά μα να έχουμε μια ενωμένη φωνή για τα θέματα αυτά περιορίζει την επιρροή μα. Πρέπει να είναι πιο αποφασιστική η ενεργειακή διπλωματία τη Ευρώπη, γιατί τα ενεργειακά μα συμφέροντα θα πρέπει να είναι μία από τι μεγαλύτερε προτεραιότητέ μα σε επίπεδο εξωτερικού εμπόριου και εξωτερική πολιτική. Χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό για να μπορέσουμε να αντισταθούμε στι πιέσει από τρίτε χώρε και να αποφύγουμε τι τρευλώσει αγορά από τρίτε χώρε που δεν σέβονται του κανόνε ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ υποστηρίζω μια ευρωπαϊκή συζήτηση που θα οδηγήσει σε μια συνένεση για να μπορέσουμε να δώσουμε μια εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να διαπραγματευτεί διεθνεί συμφωνίε εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε. Η δημιουργία τη Ενεργειακή Ένωση σημαίνει επίση καλύτερη συνεργασία με του γειτονέ μα, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερη ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των αγορών. Θέλω να τονίσω λοιπόν τη σημασία τη ενεργειακή κοινότητα για τα θέματα αυτά. Πρέπει επίση να διερευνήσουμε κοινού τρόπου αγορά φυσικού αερίου. Φυσικά θα πρέπει να σεβαστούμε του κανόνε ανταγωνισμού, του κανόνε του ΠΟΕ. Αλλά θα πρέπει, πιστεύω, να προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό και θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει το γεγονό ότι αγοράζει ενέργεια 400 δισεκατομμυρίων ω ένα πιο ισχυρό επιχείρημα. Ο πραγματικός συντονισμό σημαίνει ότι κανένα κράτο μέλο δεν πρέπει να αλλάζει το ενεργειακό του μείγμα χωρίς να έχει συντονισμό με τους γείτονε του και χωρίς να καταλάβει τι συνέπειε για του γείτονε αυτού αυτούς. Ένα περαιτέρω στοιχείο είναι η διαφοροποίηση της παροχής ε, ενέργειας σε ό,τι αφορά και τις διαδρομές και τους παρόχους ενέργειας. Θα πρέπει να εργαστούμε για τον νότιο διάδρομο για να έρθει φυσικό αέριο από την Κασπία στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με την ε, Νορβηγία, να προωθήσουμε ένα κεντρικό ε, ένα κέντρο ενέργειας για την Μεσόγειο αυτό συμπεριλαμβάνει καλύτερη συνεργασία με την Αλγερία και δημιουργία τερματικών σταθμών για υγροποιημένο φυσικό αέριο. Επίση πρέπει να έχουμε μια ανταγωνιστική και πλήρη εσωτερική αγορά. Μια πλήρη εσωτερική αγορά θα γίνει η ραχοκοκαλιά τη νέα Ενεργειακή Ένωση για την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει να αυξήσουμε τι διαμεθοριακέ ροέ ενέργεια, να έχουμε μεγαλύτερη περιφερειακή συνεργασία και μια καλύτερα συνδεδεμένη υποδομή. Θα πρέπει να βελτιώσουμε εδώ την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία, να την ενισχύσουμε και να την εφαρμόσουμε πλήρω για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να έχουμε προσιτέ τιμέ ενέργεια για τα νοικοκυριά, ιδίω για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Χρειαζόμαστε τη σωστή υποδομή για τα θέματα ενέργεια με σωστέ διασυνδέσει, ιδίω για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε την ανανεώσιμη ενέργεια στο δίκτυο ενέργεια και να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε τι νησίδε ενέργεια. Χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα διορθωτικά ταμεία, το Connecting Europe Facility, τι κοινέ επενδύσει και το μελλοντικό πακέτο επενδύσεων Juncker, ώστε να ενισχύσουμε τα σχέδια αυτά υποδομών. Τρίτο, πρέπει να μπορέσουμε να περιορίσουμε την ζήτηση ενέργειας για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας και να βελτιώσουμε την ασφάλεια ενέργειας πρέπει να μειώσουμε την συνολική ζήτηση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί όσο πρώτο, πρώτος, πιο εύκολος πόρος ενέργειας. Το καλύτερο μεγαβάτ είναι ένα μεγαβάτ που δεν καταναλώνεται ποτέ. Η ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά επέκεινα του 2020. Η βελτίωση της αποδοτικότητας δεν θα αυξήσει μοναχα την ενεργειακή ασφάλεια, θα δώσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Πλήρω υποστηρίζω την δέσμευση του κ. Γιούνκερ για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και τονίζω ότι η προτεραιότητά μα θα πρέπει να τα κτίρια, οι μεταφορέ και η παραγωγή προϊόντων τέταρτο στοιχείο είναι η μείωση του περιεχομένου άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια να μειώσουμε τι εκπομπέ αερίων θερμοκηπίου. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για τους στόχους μας του 2030 και είμαι απόλυτα προσιλωμένο στο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη αγορά για τα θέματα ανανεώσιμων ενεργειών. Ήδη το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εγκατεστημένη ικανότητα παραγωγή 44% ηλεκτρισμού από ανανεώσιμη ενέργεια. Είμαστε πρώτοι και στι τεχνολογίε ανανεώσιμη ενέργεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία μα και τη δημιουργία πάνω από 4 εκατομμυρίων πρασίνων θέσεων εργασία. Φυσικά τα κράτη-μέλη μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα να έχουν το δικό του μείγμα ενέργεια, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν προσπάθειε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε μια κοινή συμφωνία το 2015 στο Παρίσι για του στόχου αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει παίξει πρωτοπόρο ρόλο θα πρέπει να συνεχίσει να παίζει αυτό το ρόλο. Το τελευταίο στοιχείο, πέμπτο πυλώνα, είναι η έρευνα και η καινοτομία. Χρειάζονται περαιτέρω επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία και είναι κεφαλαιώδη, ιδίω για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει τι τεχνολογίε τη να φέρει αυτέ τι τεχνολογίε τη χαμηλού κόστου και χαμηλής χρήση άνθρακα, υψηλή απόδοση τεχνολογία στην αγορά. Αυτέ οι τεχνολογίε είναι απαραίτητε για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030 για κλιματική αλλαγή, για ενέργεια, οικονομικά και κοινωνικά θέματα και περαιτέρω. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα πέντε, αυτά τα πέντε βασικά στοιχεία, οι πέντε πυλώνες επί των οποίων μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανθεκτική Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση η οποία να βασίζεται με μια προορατική πολιτική για την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ του. Δεν μπορούμε να έχουμε το ένα και όχι το άλλο. Με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκομίσει καρπού και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο περιβάλλοντο και να δημιουργήσει τι θέσει εργασία που θα δώσει πράσινη ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Πριν από δύο εβδομάδε ήμουνα ενώπιον ε, τη Επιτροπή Μεταφορών για την ακρόασή μου για τι μεταφορέ και τα θέματα διαστήματο. Σήμερα προσπαθώ να κερδίσω την υποστήριξή σα για το νέο χαρτοφυλάκιο το οποίο μου δόθηκε την προηγούμενη Τετάρτη. Δεν ισχυρίζομαι ότι έγινα από τη μια μέρα στην άλλη εμπειρογνώμο στα θέματα ενέργεια. Έκανα όμω ό,τι μπορούσα για να προετοιμαστώ όσο μπορούσα καλύτερα για αυτή την ακρόαση. Και αν έχω την υποστήριξή σα, θα κάνω ό,τι μπορώ για να εξασφαλίσω ότι θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε από κοινού την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μάθω όλα αυτά που χρειάζονται για αυτά. Γιατί πιστεύω πολλά μπορούν να γίνουν σε πέντε χρόνια. Πιστεύω ότι όλοι μας το οφείλουμε στους πολίτες για να εξασφαλίσουμε ότι το όραμα μιας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ.